φορά αύριο στις 11.30. Ευχαριστώ. Και περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Είναι η έκθεση Frank Proust. καρς 2020 προς μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Το λόγο έχει ο εισηγητής Frank Proust για τέσσερα λεπτά. Ε, ε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το να σας πω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία περνάει κρίση χωρίς προηγούμενο ε, είναι γνωστό σε όλους. Ο τομέας πούλησε 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα έρετε 17 πριν την κρίση. Είναι ουσιαστικά ο... χάθηκε ο κύκλος εργασιών μιας ολοκλήρης χρονιάς. Και όμως αυτή η βιομηχανία αποτελεί πυλώνα της βιομηχανίας μας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. 23% απαιτεί πυλώνα, αποτελεί πυλώνα κοινωνικό, εμέσως και αμέσως. Είναι όμως και τεχνολογικός πυλώνας, διότι 80% των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα είναι στον τομέα της αυτοκίνητοβιομηχανίας. Βάσει όλων αυτών μπορούμε να επαναβεβαιώσουμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει θέσει την καρδιά της βιομηχανίας μας και αποτελεί και πυλώνα της οικονομίας μας εν γέννη. Όλοι ρωτώνται λοιπόν σήμερα πού πηγαίνει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Θα ήταν διανόητο, προφανώς οι αμέσως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών να μην ασχοληθούν με το θέμα. Το πράξαμε λοιπόν και με την έκθεση αυτή εξετάσαμε το σχέδιο Αυτοκινητοβιομηχανία CARS 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση εκκίνησης και ευχαριστώ προκειμένου τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για την εργασία του. Η διαδικασία CARS 2020 είναι αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων με την βιομηχανία. Παρ' όλα αυτά, έχει τα προβλήματά του το σχέδιο αυτό. Γι' αυτό και θέλουμε να προσθέσουμε εδώ την λεγόμενη προστιθέμενη αξία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την έκθεσή μου, μία φιλοδοξία έχω και μόνο, να καταθέσω καινοτόμες λύσει για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Λέω για καινοτομία γιατί έχουμε μία βραχυπρόθεσμη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε, το να βγει ο τομέας από την κρίση και μεσοπρόθεσμα βεβαίως η φιλοδοξία μας να συγκεράσουμε τις ε, πολιτικές μας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Να δώσουμε λοιπόν τη μάχη για μια Ευρώπη η οποία αναλαμβάνει δράση και η οποία κυρίως προστατεύει. Αυτό λέει η έκθεσή μου. Η οποία βασίζεται στα εξή. Πρώτον, να βελτιώσουμε την παρέμβαση της Κομισιόν με τη διατύπωση συγκεκριμένων στόχων όσον αφορά το υπερβάλλον δυναμικό παραγωγής και τον εξορθολογισμό του. Δεύτερον, με την έκθεση ζητούμε ρύθμιση με μεγαλύτερη σαφήνεια για την αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι θα γίνουν περισσότερε επενδύσει. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα η βιομηχανία, οι κατασκευαστές να βγάλουν το κεφάλι από το νερό όπω λέμε για να είναι λιγότερο ευπαθεί. Επίσης με την έκθεση υπενθυμίζουμε ότι η πρωτοπορία στον τομέα είναι το μόνο τεχνολογικό πλεονέκτημα, συγκεκριτικό πλεονέκτημα τη Ευρώπη. Α εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε να κάνουμε πολύ καλά για να μπορέσουμε με τρόπο διαρκή και βιώσιμο να προστατεύσουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Α δώσουμε περισσότερη ευελιξία στην εργασία, χάρη στον κοινωνικό διάλογο, με καλύτερε κατευθυντήριε γραμμέ, κατανοώντα και τι ανάγκε των εργοδοτών. Στούμε προκειμένου και ένα νομικό οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό τόσο εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και μεταξύ τρίτων χωρών. Από τη συνάδελφοι αυτέ είναι οι βασικέ γραμμέ τη έκθεση Αποτελεί το κείμενο συγκυρασμό των θέσεων που κατά κύριο λόγο εκφράστηκαν στην Επιτροπή. Υπερψηφίζοντα την έκθεση θα αποδείξετε ότι δεν τα βάζετε κάτω ενώπιον μια δύσκολη μάχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Χωρίς... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε αυτό το θέμα, γιατί σε σχέση με το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως, το θέμα της διαστημικής πολιτικής, ο αριθμός των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι 12 εκατομμύρια συνολικά. 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τα αυτοκίνητα. Αλλά τα τελευταία χρόνια μειώνεται αυτή η δραστηριότητα λόγω της οικονομικής κρίσης. Πέρσι πουλήθηκαν 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αλλά πριν από 5 χρόνια 17. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ελπίζω θα συνεχιστεί αυτό το σχέδιο. Πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στην Ευρώπη σε βάση μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών για τα αυτοκίνητα και μα ενδιαφέρει περισσότερο η ασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα των αυτοκινήτων. Εκεί θα πρέπει να θέσουμε την έμφαση και να είμαστε ανταγωνιστικοί εναντί του υπόλοιπου κόσμου. <coughs> Κύριο Μικολάσικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αυτοκίνητο-βιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο μας δείχνει ότι αν πρέπει να διατηρηθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το δυναμικό μας και να εστιάσουμε περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της καινοτομία για το περιβάλλον. Υπάρχει πολύ περιθώριο βελτίωσης εκεί. Η αναδιάρθρωση που αναφέρεται στην έκθεση απαιτεί την προσοχή των κρατών μελών για να υπάρξει και καλύτερος συντονισμός μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν για τις θέσεις απασχόλησης από τέτοιες πράξεις αναδιάθρωση. Πρέπει να τονίσω επίσης ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των αναδιαθρώσεων. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στο μέλλον η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να παραμείνει μια πηγή ανάπτυξης και θέσεων απασχόληση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντρές. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Σιγητά, η Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει το στόχο μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να προχωρούμε στο δρόμο της ανάκαμψης, αλλά σέρνουμε πίσω μας τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις και προβλήματα χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις που πλήττουν κυρίως τις χώρες του Νότου. Το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο θα πρέπει να κοιτάξει πέραν της κρίσης και υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες, η βελτίωση, η ανάπτυξη στην έρευνα και την ανάπτυξη, η βελτίωση εσωτερικής αγοράς, η εμπορία αυτοκινήτων πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ενώπιον των νέων προκλήσεων θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι βιομηχανικής κρίσης και επίσης τα πράσινα αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο λοιπόν είναι απαραίτητο για να μπορέσει να διατηρηθεί η αυτοκινητοβιομηχανία είναι η, ο κοινωνικός διάλογος σαν μοχλός για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπένιον. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Όσον uh, αφορά uh, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα οι το Ηνωμένο Βασίλειο, το CARS 2020 ε, ε, μπορεί να βοηθήσει την Land Rover ή την Jaguar ή παρόμοιους κατασκευαστές αυτοκινήτων για να βελτιώσουν την ε, θέση τους στην αγορά. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να βοηθηθεί η αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα στο σύνολό της έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και βεβαίως να βρεθούν οι λύσεις αυτές οι οποίες θα βοηθήσουν την αυτοκινητοβιομηχανία βιομηχανία να επιβιώσει σε έναν ε, κόσμο χωρίς διοξίδιο του άνθρακο και με λιγότερες ε, εκπομπέ. Χαίρομαι γιατί το πρόγραμμα αυτό, CARS 2020, ε, λαμβάνει υπόψη πολλά στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσει απαραίτητα και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με όλα τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθηθούν συνολικά, συνολικά ή αυτοκίνητο βιομηχανίας, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Η αυτοκινητοβιομηχανια έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση που μόλις ε, μας παρουσίασε ο κύριος Προύστ ε, ε, έχει μεγάλη αξία γιατί δείχνει ακριβώς πόσο σημαντική είναι η αυτοκινητοβιομηχανία ε, και πόσο προσφυλές θέμα αποτελεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω του σχεδίου δράσης της Οικομισιόν βεβαίως δείχνει και αυτή την ε, ε, πρόθεσή της να θέσει την αυτοκινητοβιομηχανία στην καρδιά της ανάπτυξης. Όσον αφορά το σχέδιο δράσης CARS, 2020 είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται για ένα ε, ε, πολύ καλό ε, παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να εμπνευστούμε. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο έχει βελτιώσει σημαντικά τον συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων. Πιο ευφυής νομοθεσία με τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί, πράγμα που θέλει να αποφύγει και η Κομισιόν, περαιτέρω μεγαλύτερο επιβάρυνση των, του ε, κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, θεωρεί ιδιαίτερα ε, σημαντική την διαδικασία Έγκριση τύπου ε, έτσι ώστε να ε, ε, γίνει πιο αποτελεσματική διαδικασία χωρίς να προσθέσει επιπλέον βάρος ή κόστος στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ξεκινήσει και προχωρούν πιο καθαρά αυτοκίνητα, οι εμπορικές ε, λύσεις, ε, ε, οτιδήποτε μπορεί να δώσει λύσεις στις μελλοντικές ενεργειακές προκλήσεις. Οι πράσινοι αναφέρονται στο πακέτο για την πράσινη ενέργεια. Η στρατηγική για, τις εναλλακτικές, για τα εναλλακτικά καύσιμα επίσης λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εσωτερική, μια ολοκληρωμένη αγορά για τα εναλλακτικά καύσιμα στην Ευρώπη. Όσον αφορά την έρευνα και την ε, ανάπτυξη, θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι η Κομισιόνο το 2013 παρουσίασε μία πρόταση ε, για την ε, πρωτοβουλία πράσινων αυτοκινήτων, καθαρών αυτοκινήτων σε σχέση με την ε, χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την πρόσβαση που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση μέσω του κόσμου και, η ε, Ευρωπαϊκή, και μέσω του κόσμου και μέσω των χρηματοδοτήσεων Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα προσπαθήσουμε να ε, βοηθήσουμε τις ε, εταιρείες έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ε, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε την ε, συνέχεια του ΚΑΡΣ 2020 μετά από την ε, ημερομηνία αυτή. Έχουν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και θα βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε Ρέντινγκ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας. Επόμενη σύνοδος της Ορομελίας, την 3η, 10 Δεκεμβρίου 2013, ε, από τις 8.30 μέχρι τις, 3, ε, ε, μέχρι τις 2 συγγνώμη, και ξανά